θα σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου για την εκλογή των αντιπρόεδρων. Ψήφισαν 637. Άκυρα 8. Έγκυρα 629. Η απόλυτη πλειοψηφία είναι άρα στις 315 ψήφους. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Άλβαρο 176. Αντζελίλη 241. Τζιράου 157. Κάρας 231. Μαρτίνες Μαρτίνες 257. Μακμίλαν Σκοτ 192 Παπαστάμκος 270 Πιτέλα 275 Κυρία Ποδηματά 253 Προτασιέβιτς 231 Σούριαν 203 Τάραντ 90 Βιντάλ Κουάντρας 262 Βλάζακ 184 και Βίλαντ 216 Διαπιστώνουμε πως κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε και οι 14 θέσεις αντιπροέδρων δεν ε, έχουν ακόμα καλυφθεί. Μπορείτε να ξαναδιαβάσετε αργά, παρακαλώ. Είμαστε μόνο λίγοι εδώ, αν είχα την να διαβάσετε πιο αργά. Ich Νομίζω το πρόβλημα λύθηκε. Αλλά να σας το ξαναδιαβάσω. Θα σας έλεγα τι θα γίνει από εδώ και μπρο στη διαδικασία. Επειδή λοιπόν δεν εξελέγει κανείς, θα περάσουμε σε τρίτο γύρο, αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, εδώ. Να σας πω πως τον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία και όχι απόλυτη. Αλλά απαιτείται τρίτος γύρος. Πρέπει λοιπόν να σας, ρωτήσω κυρίε και κύριοι ποιοι ε, εξακολουθούν να είναι υποψήφοι. Βεβαίω λόγω της συντριπτικής παρουσίας των υποψηφίων εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τους παρόντες. Κύριε Άλβαρο. Κύριε Αντζελίλη. Ωραία. Κύριε Αντιρό. Ευχαριστώ. Κύριος Κάρας. Κύριε Μαρτίνες Μαρτίνες. Κύριε Μακμίνα Σκότ. Κύριε Παπαστάμκο. Κύριε Πιτέλα. Κύριε Αποδηματά Κύριε Πρωτασέβιτς Κύριε Σούριαν. Κύριε Τάραντ. Θα το σκεφτώ μέχρι αύριο. Σα ευχαριστώ. Εντάξει. Κύριο κύριος Βιδαλ Κύριε Βλάζακ. Ευχαριστώ. Κύριε Βίλαντ. Ευχαριστώ. Ωραία. Okay. Με ενημερώνει η υπηρεσία πως δεν χρειάζεται νέα προθεσμία, αλλά μπορούν εάν δεν δηλώσουν ρητός πως αποσύρουν την υποψηφιότητά του, οι τωρινοί υποψήφοι να περάσουν κατευθείαν στον τρίτο γύρο. Οπότε, κύριε Τάραντ, σας ξαναρωτώ για να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω που θα είστε αύριο το πρωί νωρίς. Πόσο χρόνο έχω μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Εντάξει, κύριε Τάραντ, τότε πείτε μας μέχρι αύριο το πρωί στις 8 το εάν ε, θα είστε ακόμα υποψήφιος. Εντάξει. 7 η ώρα θα σας πάρω να σας το θυμίσω. Εντάξει. Ξέρετε, το πρωί πρωί Ωραία, λοιπόν, διακόπτη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί στις 9 για σας.